Καλησπέρα. Ας αρχίσουμε τη συνεδρίαση. Καταρχάς, συγγνώμη που χρειάστηκε να αλλάξουμε αίθουσα. Αλλά φαίνεται ότι η συνεδρίαση της ΕΝΒΙ κράτησε πολύ περισσότερο. Ελπίζω εμείς ε, να μην ε, βραδιπορήσουμε. Ελπίζω να είναι πιο σύντομη προεδρία η σημερινή θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θα ήθελα να σας θυμίσω να έχετε όλη την κάρτα ψηφοφορίας μαζί, μαζί του και αν δεν την έχετε η γραμματεία εδώ μπορεί να σας δώσει. Όλοι, όλοι είστε εντάξει, ωραία. Ωραία. Αρχίζει επισήμως η συνεδρίασή μας. Όπως ξέρετε, μοναδικό θέμα είναι η σύσταση σε σώμα του του Προεδρείου, δηλαδή να εκλέξουμε τον Πρόεδρο και τέσσερις αντιπροέδρους σύμφωνα με το άρθρο 104 του κανονισμού. Πρώτον, θα ψηφίσουμε για τον Πρόεδρο και κατόπιν θα ψηφίσουμε τους αντιπροέδρους με τη σειρά. Κάποιοι αναπληρωματικοί είναι παρόντες για να υποκαταστήσουν τακτικά μέλη. Δεν χρειάζεται τώρα να τους αναφέρω. Αλλά τέλος πάντων θα το κάνω γιατί πρέπει, το αναφέρουν οι κανόνες. Η Γκέραλντ εκπροσωπεί το Richard Κόμπετ και η Όλ Κρίστενσεν αντικαθιστά την Αγγιλέρα. Αυτά για τους σοσιαλιστές, για τους, ε, για τους σοσιαλιστές. Μιγιάν μόνο αντικαθιστά τον Άρια Σκανέτη για το ΕΛΚ. Δεν έχω άλλους αναπληρωματικούς από ό,τι ξέρω. Εντάξει. Παρακαλώ. Για την ΚΟΥΕ δεν έχω λάβει τίποτα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Α, επίσης υπάρχει κάποιος αναπληρωτής. Καλώς, καλώς, ενημερωθήκαμε. Ξέρετε ότι πάντα προσπαθούμε να διευκολύνουμε. Υπάρχει η αναγκαία απαρτία, οπότε περνάμε κατευθείαν στην ε, εκλογή του Προέδρου. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω αν υπάρχει κανείς υποψήφιος για Πρόεδρος από την πλευρά του ΕΛΚΑ. Παρακαλώ κύριος Κούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Καμπριέλ Μάτο για τη θαυμάσια προεδρία του την προηγούμενη θητεία ως αναπληρωτή συντονιστής ε, της ομάδας του ΕΛΚ έχω την ε, τιμή να προτείνω για πρόεδρο της Επιτροπής Αλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Αλέ Κάρντεκ. Άλλες προτάσεις. Όχι. Ωραία. Θεωρούμε λοιπόν ότι αναλαμβάνει την Προεδρία ο κύριος Καντέκ. Με τις προϋποθέσεις που γνωρίζετε. Ναι, ναι, ναι, ναι, αυτό κάνω. Αυτό κάνω. Λοιπόν, θα γίνει με την αναγκαία διαδικασία. Πρώτα απ' όλα ε, μου βεβαιώνουν ότι έχει υπογράψει τη δήλωση ε, συμφερόντων είναι επίσης τακτικό μέλος της Επιτροπής μας. Και το τρίτο είναι ε, αν συμφωνείτε. Συμφωνώ, ε, ρωτάω τον κύριο Καντέκ αν δέχεται την ε, θέση της Προεδρίας. Το δέχομαι, λέει ο κύριος Καντέκ. Ωραία. Και εγώ συμφωνώ, λοιπόν, εφόσον συμφωνεί ο κύριος Καντέκ, να περάσουμε, εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, μπορούμε να το κάνουμε διαβοής, όπως γίνεται συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις. Συμφωνούμε όλοι. Συμφωνούμε. Διαβοή. Ωραία. Ωραία. Να χειροκροτήσουμε για να το επιβεβαιώσουμε. Κύριε Καντέκ, παρακαλώ, σας παραχωρώ την Προεδρία. Και όλα όσα πρέπει να κάνετε ως πρόεδρος που είναι οπωσδήποτε πολλά. Και σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Ε, λοιπόν, καταρχάς σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που επιδεικνύεται στο πρόσωπό μου. Ελπίζω να είμαι στο ύψος. Θα κάνω τουλάχιστον ό,τι μπορώ. Ό,τι καλύτερο. Για να ε, μην ε, για την ψήφο σας. Σας ευχαριστώ και πάλι. Και λοιπόν τώρα, να συνεχίσουμε με την εκλογή των αντιπροέδρων. Πρώτος αντιπρόεδρος. Πρώτη αντιπροεδρία. Α, ευχαριστώ για την κάρτα μου. Πρώτη αντιπροεδρία έχουμε μία υποψήφιον. Ισαβέλα Νοβίν. Με συγχωρείτε, πρέπει, πρέπει να ρωτήσω, υπάρχει υποψήφιος ή υποψήφια. Ευχαριστώ Πρόεδρε, σας συγχαίρω για την εκλογή σας. Από πλευρά των Πρασίων και την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία προτείνω την Ιζαμπέλα Λοβίν. Ισαβέλα, δέχεστε την ε, πρόταση Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Ευχαρίστως αποδέχομαι. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Εάν δεν υπάρχουν, σας προτείνω να εκλέξουμε την Ισαμπέλα Λοβίν ως πρώτη αντιπρόεδρο διαβοήσου. Παρακαλώ να έρθει εδώ να ε, καθίσει δίπλα μου στο προεδρείο. Έχουμε ήδη το σφυρί, τον τρεπάνινο ζωάο. Λοιπόν, δεύτερη αντιπροεδρία. Υπάρχουν προτάσεις. Ευχαριστώ από πλευράς του ΕΛΚΑ. Προτείνω τον Γιαροσλάβου Αλέσα που όλοι γνωρίζετε γιατί και την προηγούμενη πενταετία ήταν ε, μέλος. Προτείνουμε τον κύριο Βαλέσα από πλευράς ΕΛΚ. Πρόεδρος. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν? Εφόσον δεν υπάρχουν,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 λοιπόν, τρίτη αντιπροεδρία. Υπάρχουν υποψήφοι. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Κύριε, παρακαλώ. Από πλευρά τη ομάδα ε, του EFD θέλω να προτείνω τον Μάρκο Φρόντε. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από πλευράς του ΕΛΚ προτείνω τον κύριο Βέρναρ Κούν. Μάλιστα. Έχουμε λοιπόν δύο υποψηφίους. Σε σύσταση σε σώμα δεν προβλέπεται συζήτηση, αλλά εάν ε, κάποιος θέλει το λόγο ένα λεπτό μπορεί να το κάνει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ συγχαρητήρια σε όλους μας. Εκτιμώ ιδιαίτερα το αξίωμα με το οποίο με επιφορτήσατε και θα συμμετάσχω με το πιο αμερόληπτο δυνατό τρόπο και ελπίζω να υπάρχει καλή συνεργασία με όλες τις πολιτικές ομάδες, όλα τα κόμματα, όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Τώρα λοιπόν, εφόσον συζητάμε για το Προεδρείο, θα ήταν καλό να σεβαστούμε τη διαδικασία για τη συνεδρίαση σύσταση σε σώμα των κοινοβουλευτικών επιτροπών. Στο άρθρο 15 του εσωτερικού κανονισμού παράγραφος 2 αναφέρεται ότι για την εκλογή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων και Κοσμητόρων θα ληφθεί υπόψη ανάγκη να υπάρξει συνολική δίκαιη εκπροσώπηση των κρατών μελών και των πολιτικών απόψεων. Όπως όλοι ξέρουμε, ως κοινοβούλιο πάντα χρησιμοποίησαμε το σύστημα DONT, ούτως ώστε να υπάρχει δίκαιη εκπροσώπηση των κρατών μελών και των πολιτικών απόψεων. Και δεν νομίζω ότι είναι σωστό η Επιτροπή μας να έχει τρία μέλη στο Προεδρείο από το ΕΛΚΑ. Το είδα να συμβαίνει πριν από μια ώρα στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπου ένα μέλος του EFDT δεν μπόρεσε να λάβει τη θέση τετάρτου αντιπροέδρου, αντιπροέδρου και στη θέση του εξελέγει κάποιο του έλπιου. Για λόγους ε, δημοκρατίας, εάν θέλουμε όντως να σεβαστούμε τις απόψεις των Ευρωπαίων πολιτών, πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις απόψεις αυτών που επικρίνουν την Ένωση. Οι απόψεις αυτές πρέπει να εκπροσωπούνται ισότιμα με όλους τους άλλους και νομίζω ότι έτσι ακριβώς θα αντιμετωπίσουμε και τις επικρίσεις κατά της Ένωσης. Κάθε υποψήφιος επιπλέον πρέπει να αντιμετωπίζεται ως άτομο και όχι μόνο ως εκπρόσωπος της ομάδας του. Και γι' αυτό θα ήθελα να ακούσω τον κύριο Αφρόντε και τον κύριο Κούν να μας παρουσιάσουν τις υποψηφιότητές τους και θα ήθελα όλοι να ακούσουμε γιατί και κατά πόσον ο κύριος Αφρόντε είναι κατάλληλος για να λάβει αυτή τη θέση. Ευχαριστώ. Ευχαριστή Ζαβέλα. Όχι, όχι. Δεν θα ξεκινήσουμε συζήτηση τώρα. Θα συμβαστούμε τους δημοκρατικούς κανόνες μέσω της ψηφοφορίας. Δεν μπορείτε εκ των υστέρων να κάνετε αφισβητήσεις, θα σεβαστούμε τους δημοκρατικούς κανόνες, θα περάσουμε στην ψηφοφορία. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία προτείνουμε να ψηφίσουμε πρώτα για τον κύριο Αφρόντε. Παρακαλώ πατήστε το πράσινο κουμπί αν θέλετε ο κύριος ε, Αφρόντε να εκλεγεί αντιπρόεδρος και αν θέλετε ο κύριο Κούν σας παρακαλώ να πατήσετε το κόκκινο. Θέλετε να κάνουμε πρώτα ένα τεστ. Εντάξει, είστε όλοι έτοιμοι να ψηφίσετε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Εντάξει. Βάλετε στη σχισμή την κάρτα σας. Αν θέλετε να ψηφίσετε τον κύριο Αφρόντε πράσινο, κουν κόκκινο. Βάσει των δημοκρατικών κανόνων. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρχεται. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 11 ψήφοι υπέρ του κυρίου Κούν και 9 υπέρ του κυρίου Αφρόντα. Δεν είναι απόλυτη πλειοψηφία, πρέπει, γιατί υπάρχουν και δύο αποχές. Θα πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. Μηδενίστε παρακαλώ το μηχάνημα, παρακαλώ ξαναψηφίστε. Άρχεται. Le vote est fermé. Πέρας Δώδεκα για τον κύριο Κούν, εννέα για τον κύριο Αφρόντε. Εκλέγεται τρίτος αντιπρόεδρος ο κύριος Κούν. Je Διευκρινίζω ότι ο κύριος Αφρόντε θα συμμετάσχει προφανώς ενεργώς στις εργασίες μας. μιλάτε για δημοκρατία, αλλά δημοκρατία στην Αγγλία σημαίνει ότι επιτρέπεται ο κόσμος να παίρνει το λόγο. Κανένας από τους υποψήφιους δεν έλαβε το λόγο. Ε, μάλλον για ευρωπαϊκή δημοκρατία μου μοιάζει αυτό που δεν είναι αγγλική δημοκρατία, που δεν είναι αληθινή δημοκρατία. Ε, Αυτοί είναι οι κανόνες. Ε, δεν θα ξεκινήσουμε συζήτηση. Δεν θα ξεκινήσουμε παρακαλώ συζήτηση. Α, περάσουμε τώρα στην εκλογή του Δετάρτου Αντιπροέδρου. Υπάρχουν υποψήφοι. Υποψήφοι για την ε, θέση του Τετάρτου του Προέδρου. Ε, ε, ναι, η πολιτική μου ομάδα προτείνει την κυρία Ρενάτα Μπριάνκο. Υπάρχουν άλλες υποψηφιότητες. Όχι προτείνω να εκλέξουμε την κυρία Οριάνκο Βριάνο διαβοής. Merci. Le bureau... Ευχαριστώ. Ωραία. Συμπληρώθηκαν οι θέσει του Προεδρείου. Επόμενη συνεδρίαση στις 22 του μηνός. Θα δούμε και με τη γραμματεία. Αλλά προτείνω ή δυνατόν συνεδρίαση να γίνει από τις 2 και όχι από τις 9 το πρωί. Γιατί να μην ξεχνάτε ότι στις 21 δεν είναι αργία και είναι όλα κλειστά. Θα δούμε. Αλλιώς στις 23, 9 το πρωί. εσείς δεν πιστεύετε στη δημοκρατία, ποτέ σας αγνοώ. Ε, Καλό απόγευμα, κυρία μου. Λοιπόν, για τη συνεδρίαση θα γίνει στις 22, στις 2 το μεσημέρι. Ή αυτό ή καθόλου. Θα οργανωθούμε λοιπόν και θα σας ενημερώσουμε μέσω mail για την ακριβή ώρα της συνεδρίασης στις 22. Ευχαριστώ. Και καλό απόγευμα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.